Επαναλαμβάνεται η συνεδρία. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι έκθεση Wolf Klintz με θέμα του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον αφορά ορισμένου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητέ αξίε. Ο κύριο Κλίντ, εισηγητή, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τον Ιούλιο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την πρότασή της